panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. επαναλαμβάνεται η συνεδρία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Χαιρετίζω τα μέλη που είναι παρόντα και τον κύριο Επίτροπο. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίασης έχουν ε, διανεμηθεί. Έχετε κάποια σχόλια σε σχέση με τα πρακτικά. Εάν όχι, θεωρούνται τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί. Ερχόμαστε στο επόμενο λοιπόν σημείο της ε, διάταξης, τη δήλωση της Κομισιόν